Αγαπητοί συνάδελφοι, καλώ ήρθατε στι ψηφοφορίε. Ξεκινάμε με την έκθεση του συναδέλφου Βαλκάρ Σελσίσο. Καθίστε σιγά σιγά. Έχουμε ονομαστική ψηφοφορία. Συνάδελφος Ντάρτμουντ. Κύριε Πρόεδρε, θέλω να ρωτήσω αν μπορούμε να συγχαρούμε τον πρώην Πρόεδρο της Επιτροπής, τον κύριο Μπαρόζο, για το διορισμό του στην Golden Sachs. Επίσης, θέλω να εκφράσω και την ανησυχία μου, διότι η σύνταξή του ως πρώην πρόεδρος της Επιτροπής δεν του αρκεί. Δεν ξέρω αν